please. going to start. Παρακαλώ, θα ξεκινήσουμε την συνεδρίαση. Σας καλώ να πάρετε θέσεις. Με μεγάλη χαρά Κυρίσω την άναξη της πρώτης συνεδρίασης της Επιτροπής ΕΝΒΗ. Θα ξεκινήσουμε μια ανταλλαγή απόψεων με τον ε, Υπουργό, τον κύριο Λέπα, τον Υπουργό Γεωργίας και Δασοκομείας. Χαιρόμαστε που είστε εδώ μαζί μας σήμερα. Έχουμε μια μισή ώρα περίπου μπροστά μας για να είμαστε βέβαιοι ότι όλοι οι ευρωβουλευτές που θέλουν να πάρουν το λόγο θα μπορέσουν να παρέμβουν. Θα είμαι κάπως σκληρός, ε, αυστηρός έτσι, στα θέματα τα χρονικά. Δύο λεπτά για τους συντονιστές, ένα λεπτό για τους υπόλοιπους ευρωβουλευτές. Όταν θα, ξεπερνάμε, θα ξεπερνάει κάποιος αυτό το όριο, θα σας διακόπτω και θα δίνω το λόγο στον επόμενο ομιλητή. Δεν θα διστάσω δηλαδή να, να σας αναγκάσω να σεβαστείτε τον χρόνο. Λοιπόν, έχετε το λόγο κύριε Υπουργέ. Arvoisa herra puheenjohtaja, hyvät Euroopan parlamentin ympäristö- Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας, Διατροφικής Ασφάλειας, κυρίες και κύριοι, είναι χαρά μου που είμαι ο πρώτος υπουργός που θα μιλήσει στην Επιτροπή αυτή. Το Κοινοβούλιο εκπροσωπεί τους Ευρωπαίους πολίτες. Είναι ένα πολύ σημαντικό όργανο και βεβαίως ε, προασπίζει τις ευρωπαϊκές αξίες. Είναι μια σημαντική ευκαιρία ε, έτσι, για να έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων μεταξύ θεσμικών οργάνων. Θα ήθελα να σας συγχαρώ καταρχήν για την εκλογή σας ε, στο Κοινοβούλιο και αυτή την Επιτροπή. Η Επιτροπή αυτή ε, παίζει ένα σημαντικό ρόλο. Παρακολουθώ με μεγάλο ενδιαφέρον το πώς ξεκινάτε τις εργασίες σας. Η Φιλανδική Προεδρία έχει αναλάβει εδώ και τρεις εβδομάδες και μπορώ να σας πω με μεγάλη χαρά ε, ποιες είναι οι προ... πολιτικές προτεραιότητες της Προεδρίας μας και να απαντήσω και σε όποιες ερωτήσεις έχετε. Πολλά πράγματα έχουν αλλάξει από την προηγούμενη Προεδρία μας. Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μετά τη συνδίκη της Λισαβόνας έχει ενισχύθει καθώς και ο ρόλος της Προεδρίας έχει αλλάξει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, οι υπηρεσίε Εξωτερική Δράση έχουν πλέον του δικού του εκπροσώπου στα όργανα. Οι προτεραιότητέ μα κατά τη διάρκεια τη Προεδρία μα έχουν να κάνουν με την αντιμετώπιση τη κλιματική αλλαγή, η προώθηση των κοινών θεμελιωδών αξιών τη Ένωση και του κράτου δικαίου, η ενίσχυση τη ασφάλεια και η ενίσχυση μιας ε, ε, της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινωνικής Συνοχής. Έχουμε λοιπόν σημαντικού φακέλου να αντιμετωπίσουμε το επόμενο εξάμεινο. Προσπαθούμε να βρούμε λύσει σε ό,τι αφορά το στο νομικό πλαίσιο, που είναι ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα που θα απασχολήσουν την Προεδρία μα. Επίση, θα προσπαθήσουμε να φτάσουμε σε συμφωνία για τη μακροπρόθεσμη στρατηγική για το κλίμα ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να δράσει αποφασιστικά για να επιτευχθούν οι στόχοι των Παρισίων έτσι ώστε να μπορέσουμε να περιορίσουμε την υπερθέρμανση στον 1,5 βαθμό Κελσίου. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να φτάσουμε σε μηδενικές εκπομπές έως το 2050. Θα ζητήσουμε επίσης και, να μιλήσουμε επίσης για τη βιοπικιλότητα και προσπαθήσουμε να μειώσουμε την έλλειψη, την απώλεια βιοποικιλότητας. θα πρέπει να δεσμευτούμε ε, στην προσπάθεια για το τι θα συμβεί μετά το 2020 σε ό,τι αφορά ε, τα ζητήματα βιοπικιλότητας στο Υπουργείο Γεωργίας και Αλίας ένα βασικό ζήτημα θα είναι η μεταρρύθμιση της κοινωνικής πολιτικής θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να φτάσουμε σε κοινή θέση στο Συμβούλιο επ' αυτού. Η μεταρρύθμιση τη κοινωνική πολιτική συνδέεται στενά βεβαίω με την πρόοδο ε, στι διαπραγματεύσει για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Επιπλέον, η άτυπη Υπουργική Σύνοδο στο Ελσίνκι το Σεπτέμβριο ε, έχει να κάνει με, την, ε, ε, με τον άνθρακα στον τομέα της γεωργίας η δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα. Θα πρέπει να σημειωθεί, προ, να σημειωθεί πρόοδος και στο ζήτημα του Ταμείου Αλίας και του Ταμείου Θαλάσσης. Το θέμα των ΤΑΚ επίσης στον τομέα της Αλίας θα πρέπει να επιληθεί. Εμείς ε, ακολουθούμε βεβαίως ε, τις αρχές της του ανοιχτού χαρακτήρα ε, της, ε, σωστής διακυβέρνησης και βεβαίως της βιώσιμης διακυβέρνησης. Ε, είναι 500.000 ευρώ το κόστος από τις μετακινήσεις λόγω των συνεδριάσεων. Θα περιώσουμε τις συνεδριάσεις λοιπόν αυτές και θα διασώσουμε τα χρήματα αυτά σε διάφορα project στην Ουγκάντα, στο Λάο, στη Βιρμανία, ε, στο Βιετνάμ, συγγνώμη. Ε, είναι διατομεακά τα ζητήματα του περιβάλλοντος, είναι οριζόντια. Δεν μπορούν να βρεθούν λύσεις σε συγκεκριμένου τομεί για το θέμα του περιβάλλοντο. Και οι όποιε λύσει βρίσκονται επηρεάζουν όλου του τομεί. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται μια ευρεία διαθεσμική και διατομεακή συνεργασία. Και οι πολιτικέ γεωργία και αλλία πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τι λοιπέ πολιτικέ. Θα ήθελα να αναφερθώ τώρα σε κάποιε προτεραιότητε που έχουν να κάνουν με τι αρμοδιότητε τη δική σα επιτροπή ε, και όπου θα θέλαμε να σημειώσουμε πρόοδο κατά τη διάρκεια τη Προεδρία μα. Πρώτα απ' όλα η μεταρρύθμιση της κοινωνικής πολιτικής. Όπως είπα, θέλουμε να σημειώσουμε όσο γίνεται μεγαλύτερη πρόοδο στο θέμα αυτό της μεταρρύθμισης, της ΚΑΠ. Εάν προχωρήσει το πολιτισμο νομικό πλαίσιο, θα μπορέσουμε να φτάσουμε και σε γενική συμφωνία στο Συμβούλιο. Χαίρομαι που τα κράτη-μέλη στο Συμβούλιο δεσμεύτηκαν ε, για φιλόδοξους στόχους σε ό,τι φορά τα κλιματικά και περιβαλλοντικά ζητήματα. Ένα υγιές περιβάλλον, ένα καλύτερο κλίμα, μια καλύτερη ε, χρήση, πιο βιώσιμη χρήση ε, των πόρων μας ε, είναι απαραίτητα στοιχεία για την επιβίωσή μας αλλά και για τον τομέα της γεωργίας. Η νέα δομή τη γεωργική πολιτική θα καταστήσει υποχρεωτικά κάποια περιβαλλοντικά μέτρα και θα δώσει στα κράτη-μέλη τη δυνατότητα να θεσπίσουν και εθνικά περιβαλλοντικά μέτρα στα πλαίσια του πρώτου και του δεύτερου πυλώνα. Οι διαπραγματεύσει ε, όμω είναι ακόμα εν εξελίξη. Ω εκπρόσωπο τη Προεδρία πρέπει να σα πω ότι η νέα πράσινη αυτή αρχιτεκτονική περιλαμβάνει υπόψη, λαμβάνει υπόψη ε, τι διαφορετικέ ανάγκε και ιδιαιτερότητε τη κάθε χώρα και τη κάθε περιφέρεια. Γι' αυτό θέλουμε να πάρουμε μέτρα περιβαλλοντικά και κλιματικά χρήσιμα, χρήσιμα και στοχευμένα. Θα πρέπει να υπάρχει λοιπόν ισορροπία στους στόχους αυτούς. Να πω τώρα δύο λόγια για τα δάση. Ένα ζήτημα στο οποίο θα ήθελα να την προσοχή σας είναι η παγκόσμια αποψήλωση ε, η οποία προχωράει με γιγάντιους ρυθμούς και όταν μιλάμε για εξαφάνιση των δασών πρέπει να δούμε την ευρύτερη εικόνα διότι οι βιώσιμες λύσεις ε, σημαίνει ότι πρέπει και εδώ να παρεύουμε σε πολλούς τομείς για να μπορέσουμε ε, να προωθήσουμε την αναδάσωση. Χρειαζόμαστε βιώσιμη διαχείριση των δασών και, και προστασία των δασών. Πρέπει επίσης ε, τα δάση τα οποία έχουν ε, πληγεί, τα οποία έχουν υποστεί ζημιά, να μπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους. Κατά τη της Προεδρίας μας είμαστε διατεθειμένοι να προωθήσουμε μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματο τη αποψήλωση. Τώρα, να πω τη λόγια για τη συμφωνία με το Μερκοσούρ. Πριν από ένα μήνα περίπου φτάσαμε σε πολιτική συμφωνία, εμπορική συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Μερκοσούρ. Πολύ σημαντική αυτή η εμπορική συμφωνία. Το ότι φτάσαμε σε αυτό το αποτέλεσμα με την παρούσα πολιτική συγκυρία δεν ήταν καθόλου ε, προφανές. Βεβαίω στον τομέα τη γεωργία υπάρχουν ανησυχίε ε, και για τα γεωργικά προϊόντα αλλά και για ζητήματα βιωσιμότητα. Το αντιλαμβάνομαι αυτέ τι ανησυχίε. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό μάλιστα η συμφωνία του Μερκοσούρ να περιλαμβάνει, περιλαμβάνει ήδη μάλλον ένα κεφάλαιο για τη βιωσιμότητα. Η συμφωνία των Παρισίων και η αρχή τη προφύλαξη περιλαμβάνονται και αυτά τα στοιχεία στη συμφωνία με το Μερκοσούρ. Όταν λοιπόν θα εφαρμοστεί αυτή η συμφωνία, όταν θα υλοποιηθεί, θα πρέπει οι αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης να γίνουν σεβαστές και οι προϋποθέσεις οι εμπορικές να είναι ικανοποιητικές και για τις δύο πλευρές. Το Μερκοσούρ, ε, όπως και στις άλλες εμπορικές συμφωνίες, υπάρχουν αυτές οι ρήτρε ε, για να υπάρχει εμπιστοσύνη και του καταναλωτή σε ό,τι αφορά τη διατροφική ασφάλεια, επίσης η φυτοκοινωνική ε, κατάσταση, η προστασία των ζώων και αυτά δεν πρέπει να διακυβευθούν. Ακούσαμε την ανακοίνωση της Κομισιόν την περασμένη εβδομάδα για τη μεταφορά ζώων ε, σε μεγάλες αποστάσεις, ζωντανών ζώων. Μιλάμε για μεγάλες αποστάσεις, σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες συχνά. Ε, και βεβαίως εδώ ξεπερνάμε συχνά τα, τα όρια του αποδεκτού, ε, συχνά σε κλειστά κοντέινερ, όπου οι απαιτήσει, οι προδιαγραφές δεν πληρώνται. Ε, για μας είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό και χαιρόμαστε που η Κομισιόν το ανέφερε την περασμένη εβδομάδα. Υπάρχει και ένα ζήτημα προστασίας του καταναλωτή εδώ. Ο καταναλωτής πρέπει να γνωρίζει ότι η όλη αλυσίδα παραγωγής είναι υπεύθυνη, επιδεικνύει επιθυνότητα και ότι η ευημερία των ζώων γίνεται σεβαστή σε όλη τη διάρκεια της αλυσίδας αυτής. Αυτό ισχύει και για τα ζώα εκείνα τα οποία εξάγονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλος, θα ήθελα να πω δύο λόγια για την μικροβιακή αντίσταση. Είναι μια εξαιρετικά σημαντική παγκόσμια απειλή για την ανθρώπινη υγεία και για την υγεία των ζώων, αλλά και για, την, για το περιβάλλον και τη διατροφική ασφάλεια. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ενεργή του ε, δράση για το θέμα αυτό. Μπορεί να έχει αλλάξει βεβαίω η σύνθεση στην Επιτροπή σας, αλλά το θέμα παραμένει επίκαιρο. επίκαιρο. Πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέκρινε ένα κανονισμό για τα κτηνιατρικά φάρμακα που απαγορεύει την χρήση αντιβιωτικών με αυξητική ε, ε με αυξητικό αποτέλεσμα. Ε, είναι πολύ σημαντικό να μειωθεί η χρήση των αντιβιωτικών ε, για να είναι και πιο αποτελεσματική η χρήση τους. Η χρήση των αντιβιωτικών μπορεί να μειωθεί εφόσον επενδύσουμε στην ευημερία των ζώων και στην υγεία των ζώων. Πρέπει η χρήση των αντιβιωτικών να ελέγχεται, να ε, βασίζεται σε συγκεκριμένα επιστημονικά στοιχεία. Χρειάζεται αποφασιστικότητα από όλου του εμπλεκόμενου φορεί και από τι ε, δημόσιε διοικήσει. Χαίρομαι που υπάρχει συνεργασία ε, στον τομέα της υγείας από διάφορους τομείς, ε, μια συνεργασία που λειτουργεί αποτελεσματικά. Η αντιμετώπιση της μικροβιακής αντοχής χρήζει παγκόσμιας συνεργασίας και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι στην πρώτη γραμμή και να, δείξει δείχνει το δρόμο. Αξιότιμα μέλη της Επιτροπής, Κύριε Πρόεδρε, είναι πολυσχηδή όλα τα προβλήματα αυτά στα οποία αναφέρθηκα. Ως πρόεδρος στο Συμβούλιο Γεωργίας και Αλίας, εγώ πρέπει να προσπίσω την διατροφική ασφάλεια μεταξύ άλλων. Θα πετύχουμε λοιπόν το καλύτερο αποτέλεσμα εφόσον λάβουμε υπόψη μας τη βιωσιμότητα των θεσμών μας και να συνεργαστούμε και συνεργαστούμε με όλους τους αρμόδιους φορείς. Ελπίζω να μπορέσουμε να σημειώσουμε πρόοδο στην Προεδρία μας. Εμείς εργαζόμαστε ένα πνεύμα συνεργασίας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Υπουργέ. Υπάρχουν πολύ σημαντικά στήματα όπως είναι η κοινωνική πολιτική, η πολιτική συμφωνία με τις χώρες Μερκοσούρ και άλλα θέματα στα οποία αναφερθήκατε. Θα έχουμε την ευκαιρία να έχουν μια ανταλλαγή απόψεων με τρεις υπουργούς της Φιλανδία σήμερα και αύριο και έτσι θα αποκομίσουμε μια συνολική εικόνα για τους στόχους της Προεδρίας σας. Και αυτό να το έχουμε υπόψη, είναι σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό δηλαδή να έχουμε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων όλοι μαζί με τους εκπροσώπους της Φιλανδικής Προεδρίας, γιατί στο Στρασβούργο που ακούσαμε τον Πρωθυπουργό σας και εδώ που σας ακούμε σήμερα βλέπουμε ότι στο προσκήνιο βρίσκονται περιβαλλοντικοί στόχοι για την Προεδρία σας. Άρα θα υπάρχει μια πολύ καλή σχέση και ατμόσφαιρα και μας χαροποιούν οι προτεραιότητες που ακούμε διαστόματό σας. Τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στους ε, συντονιστές ή τους εκπροσώπους αυτών, όπως επελέξαν από τις πολιτικές ομάδες. Να σας πενθυμίσω τον κανόνα, εφόσον αυτή είναι η πρώτη τακτική μας συνεδρίαση, κάθε συντονιστής έχει στη διάθεσή του δύο λεπτά για να θέσει τις ερωτήσεις του. Και ε, όταν ολοκληρωθεί ο πρώτος γύρος, με τους συντονιστές. Θα λάβετε ξανά κύριε Υπουργέ το λόγο για να απαντήσετε. Να ξεκινήσουμε με το ΕΛΚ λοιπόν. Τζέσικα Πορφιάτ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κίτος κύριε Υπουργέ Λέπα για την παρέμβασή σας και τις προτεραιότητες που αναφέρατε. Φιλανδία και Σουηδία έχουν μακρά ιστορία βιώσιμης ε, ε, ανάπτυξης και προστασίας των δασών, κάτι για το οποίο είμαστε υπερήφανοι. Η ενεργός διαχείριση των δασών ε, μας βοηθά άλλωστε να πετύχουν και τους περιβαλλοντικούς στόχους. Δεν υπάρχει αμφιβολία για το πόσο σημαντικά είναι τα δάση για το κλίμα. Και αν έχουμε καλή διαχείριση και με τη δέσμευση του, του άνθρακα και τα καλά πρώτα ξύλια, μπορούμε να αξιοποιούμε όλο τον κύκλο ζωής των δασών. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα ε, ανανεώσιμα υλικά, να προωθήσουμε την βιοοικονομία με χαμηλότερες εκπομπές οξυδιού του άνθρακα. Τι θα κάνετε εσείς για να ε, διασφαλίσετε τις εθνικές αρμοδιότητες στον τομέα της δασοκομείας στη διάρκεια της Προεδρίας σας. Αυτό είναι το ερώτημά μου πώς θα προωθήσετε τη βιώσιμη αυτή, η το βιώσιμο αυτό κλάδο. Σας ευχαριστώ και πάλι και προσβλέπω σε μια επικοδομητική συνεργασία μαζί σας. Κάθε επιτυχία στο έργο σας. Προεδρο. Uh, Πρόεδρος, βάλατε ψηλά τον πίσω ότι αφορά το κλίμα. Από τους ε, συντονιστές ε, Σαλντεμόζε εκ μέρους των συντονιστών. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς θέλω να σας καλωσορίσω και να σας πω ευχαριστώ εκ μέρους ομάδας μας Σοσιαλιστών και Δημοκρατών ε, που αναφέρατε ως προτεραιότητα το κλίμα και την ε, βιωσιμότητα. Πολύ σημαντική στόχη και νομίζω ότι θα έχουμε πολύ καλή συνεργασία. Όπως γνωρίζετε, και ως Προεδρία στις τελευταίες θητείες ε, η Κομισιόν ε, κυρίως ενδιαφέρθηκε και εργάστηκε για να υπάρχει διαφάνεια στη διαδικασία έγκρισης των φαρμάκων. Δεν είναι δική σα αρμοδιότητα να καταθέσετε νέα νομοθεσία. Απλά ερωτώ, αναγνωρίζετε ότι δεν υπάρχει επαρκή ανεξαρτησία ε, σε Ευρωπαϊκή Ένωση ότι αφορά την έγκριση φυτοφαρμάκων. Δηλαδή πιστεύετε ότι πρέπει να δοθούν περισσότερα μέσα στην ΕΣΑ στον, ε, ή στον Οργανισμό Χημικών Προϊόντων για να διενεργούν τις δικές τους μελέτες και να μπορούν να ασκούν περισσότερες πιέσεις και να διατυπώνουν περισσότερες υποδείξεις και συστάσεις. Και σε ό,τι αφορά και τη διαχείριση των δασών, σε συνέχεια της προηγούμενης παρέμβασης, θεωρώ ότι η αηφορία, η βιωσιμότητα θα μας δώσει τη δυνατότητα εν μέρη να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις του κλίματος. Τι θα κάνετε όμως ε, ώστε να γίνουν σεβαστοί οι κανόνες που ήδη υφίστανται από όλα τα κράτη-μέλη. Υπάρχουν χώρες οι οποίες εισάγουν παράνομη ξυλία εντός Ένωσης. Πώς θα διασφαλίσετε την εφαρμογή της νομοθεσίας. Γιατί είναι και δική σας αρμοδιότητα ο σεβασμό, δηλαδή η επιτήρηση του σεβασμού της νομοθεσίας. Σας ευχαριστώ εκ μέρους της ομάδας μου για την ε, συνεργασία μας εκ των προτέρων. Σα Σας ευχαριστώ πολύ και τώρα περνάμε στην ομάδα Renew. Νίλς Τόρβαλς. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε ε, Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω, να καλωσορίσω και τον Υπουργό στην ωραία μας παρέα. Η ε, συζήτηση βεβαίως ε, είναι πολύ ενδιαφέρουσα και φυσικά όμως δεν μπορεί κανείς μέσα σε δύο λεπτά να πει κανείς αυτά που θέλει ε, και πρέπει να σας πω ότι κάθε λεπτό που περνάει ε, ε, βλέπουμε να, λιώνει, να λιώνουν λίγο περισσότερο οι πάγοι, βλέπουμε να έχουμε λιγότερα ψάρια στους ωκεανούς μας και αυτά. Εν πάση περιπτώσει όμως αυτά δεν μας αφορούν σήμερα εδώ και ούτως ή άλλως και η Φιλανδία και όλες οι γύρω χώρες πρέπει να ε, προχωρήσουν. Tota, ε, Μα είπατε προηγουμένω ε, για την δέσμευση του άνθρακα, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει με τις παραδοσιακές μορφέ της γεωργίας. Θα ήταν καλό λοιπόν να μας πείτε τι, θε, τι προτίθεται να κάνει η ε, Φιλανδία όσον αφορά τη γεωργία σε σχέση με τη δέσμευση και αποθήκευση του άνθρακα και ποιε θα είναι οι προτεραιότητε τη θα είναι δηλαδή δηλαδή οι προτεραιότητες στη διάρκεια της εξάμηνης προεδρίας. Πράσινη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ για την ε, παρουσία σας, λέει ο κύριος Ζαντό. Ε, ε, νομίζω ότι είναι ενδιαφέρον να συζητήσουμε για όλα αυτά. Ε, πάντως θα ήθελα να μου πείτε το εξής ε, ε, στην, ε, στα συμπεράσματα της η Κομισιόν αναφέρεται και στην αποψήλεση. Ξέρετε όμως κύριε Υπουργέ ότι εκατομμύρια εκτάρια λόγω της, των εισαγωγών μας σε κακάο, σε διάφορα άλλα όπως το φινικέλαιο και άλλα προϊόντα έχουν σαν αποτέλεσμα την αποψήλωση χιλιάδων εκταρίων. Τι θα κάνετε γι' αυτό επίσης ε, διατίθεστε ευνοϊκά ε, να εισαχθεί ε, στην νομοθεσία, στην ευρωπαϊκή νομοθεσία, δεσμευτική νομοθεσία σχετικά με τις επιχειρήσεις οι οποίες είτε συμμετέχουν είτε όχι στην αποψήλωση και ε, και όσον αφορά ε, λοιπόν την ε, αλυσίδα προμήθειας προϊόντων γεωργικών και δασοκομείας να εφαρμοστούν όλα τα, όλες οι αποφάσεις αυτές όσον αφορά το Mercosur. Καταλαβαίνω αυτά που λέτε γιατί μας είπατε ότι υπάρχει και ένα κεφάλαιο για την ανάπτυξη αλλά ξέρετε αυτό το κεφάλαιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη δεν πρόκειται να λύσει τίποτα όπως λέτε εσείς και διατείνεστε εσείς, γιατί δεν υπάρχει καμία υποχρεωτική ενέργεια. Ξέρετε, όπως και, εγώ γνωρίζω πολύ καλά, ότι ε, με, την, με τον Μπολσενάρο στην ηγεσία της ε, χώρας, στη Βραζιλία έχει προχωρήσει με μεγάλη ταχύτητα η αποψήλωση και επίσης η πολιτική του Μπολσενάρο ε, είναι απολύτως αντίθετη με οποιαδήποτε δέσμευση είχε ληφθεί στα πλαίσια της συμφωνίας Μερκοπού, Μερκοσούρα από από τη στιγμή λοιπόν που η Κομισιόν θέλει από ό,τι λέει να εξισορροπήσει την κατάσταση, τι θα κάνετε έτσι ώστε να σταματήσει η αποψήλωση στην Αμαζονία. ID, ομάδα ID, επόμενος ομιλητής. Κύριος ε, Χάκα Ράινεν. Κύριε Υπουργέ, να σας ευχαριστήσω γιατί αναφερθήκατε εδώ στο θέμα των δασών. Η Φιλανδία επενδύει στην δασοπονία καθώς επίσης και στη διαχείριση των δασών εδώ και πολλά χρόνια. Τώρα ε, τα δάση, το πρόβλημα με τα δάση ε, μεγαλώνει όπως και το θέμα των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακος. Είχαμε πολλές δασικές πυρκαγιές, παρόλα αυτά κάθε φορά βλέπουμε ότι αναγεννάται το δάσος. Ο Καναδάς είναι η δεύτερη, πιο, η δεύτερη χώρα με, τις, ε, με, τα, με τη μεγαλύτερη ε, ποσότητα και αριθμό κονοφόρων ε, δέντρων και έχουν δημιουργήσει τέτοιες λεκάνες αποθήκευσης ε, διοξιδίου του ε, άνθρακος. Κάτι αντίστοιχο ε, θα μπορούσαμε να κάνουμε και στη Φιλανδία, μια και υπάρχει η τεχνογνωσία και η απαραίτητη τεχνολογία, η βιωσιμότητα δεν πρέπει να εξαρτάται από τις εισαγωγές όπως μπορεί να συμβαίνει σε άλλους τομείς. Επιπροσθέτως, ε, μέσω των ε, δασών ε, μπορεί να παραχθεί ανανεώσιμη ενέργεια. Η χρήση των δασών όμως έχει φτάσει στο μέγιστο σημείο και χρησιμοποιούμε τεράστιες ποσότητες ε, ε, δασικών προϊόντων και ξυλίας ε, το χρόνο που σημαίνει ότι δεν θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση της δημιουργίας λεκάνων αποθήκευσης. Το έχει λάβει υπόψη του αυτό ο κύριος Υπουργός, η Άννα Βιαλεύσκα. ECR. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητέ Πρόεδρε, Αξιότιμη Υπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι, άκουσα τους φιλόδοξους στόχους της χώρας σας, κύριε Υπουργέ. Δύσκολη καιρή όμως, διότι έχουμε να διαπραγματευτούμε τον προπολογισμό, που δεν έχει εγκριθεί ακόμη. Πρόκειται για έναν προπολογισμό που βλέπουμε χαρακτηρίζεται από όλο και λιγότερους πόρους για την κοινή πολιτική και από ε, μεγάλες ε, περικοπές για την ε, πολιτική αυτή. Πώς θα διαπραγματευτείτε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα διάφορα κράτη-μέλη. Σύντομα θα συγκροτηθεί η νέα Επιτροπή της Ένωσης. Πώς θα εξασφαλίσετε περισσότερα χρήματα για την κυνηγιορική πολιτική. Δεύτερο ερώτημα. Πώς θα αντιμετωπίσετε το πρόβλημα των ανισοτήτων μεταξύ των αγροτών, που θεωρώ ότι θα πρέπει να παίρνουν ε, τα ίδια χρήματα. Επίσης, ε, μείωση της γραφειοκρατίας ε, του διοικητικού άχθους. Πώς θα σταματήσουν να υπάρχουν αυτές οι συμφορήσεις στον πρώτο πυλώνα κυρίω. Είναι ένα θέμα που δημιουργεί πολλά προβλήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και νομίζω ότι χρήζει της προσοχής σας. Αναφερθήκατε και στην περιοχή Μερκοσούρ. Πρόκειται για χώρες συνδεδεμένες ε, με την Ένωση. Σύντομα, φαντάζομαι ότι θα έχετε νέα από τους αγρότες, γιατί εμάς τουλάχιστον ε, μας ε, μιλούν οι αγρότες και μας εκφράζουν τις ανησυχίες τους για την ασφάλεια των τροφίμων. Τα δικά μας πρότυπα στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων είναι πάρα πολύ αυστηρά. Όμως ε, το Μερκοσούρ υπολείπεται σε πολύ μεγάλο βαθμό σε ό,τι αφορά αυτά τα πρότυπα. Ωραία, υπεγράφει τη συμφωνία και μετά τι μελγενέστε. Αυτό είναι το ερώτημά μου. Πρέπει να είμαστε αυστηροί για το σεβασμό των ε, προτύπων και κανόνων ασφάλειας τροφίμων. Τελευταίο ερώτημα. Είστε ε, ένα καλό παράδειγμα για τη διαχείριση των δασών. Θα προετοιμάσετε μήπως μια εργαλειοθήκη, ένα, ε, μια μεθοδολογία, ώστε να μπορούν να βρουν μιμητές ε, σε άλλες χώρες τα όσα κάνετε εσείς. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Ψήλβια από την ΚΟΕ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, κύριε Λέπα, ε, χαίρομαι ιδιαίτερα που η Φιλανδία έθεσε το θέμα της κλιματικής αλλαγής ως προτεραιότητα της Προεδρίας της και που θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι στην πρώτη γραμμή. Αναφερθήκατε στη Γεωργία όμως στην ομιλία σας. Είναι κάτι που δεν το συζητούμε επαρκώς. Μιλάμε συνέχεια για τη μείωση των εκπομπών. Ναι, αλλά πρέπει επίσης να ενισχύσουμε και την ε, δυνατότητα δέσμευσης άνθρακα. Ε, πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Ποιες είναι συγκεκριμένες προτάσεις δηλαδή προς την κατεύθυνση αυτή. Προς τους γεωργούς. Πώς μπορούμε να καταστήσουμε τη γεωργία περιβαλλοντικώς βιώσιμη στα πλαίσια και της, της μεταρρύθμισης της κοινής πολιτικής. Και ένα ακόμα ερώτημα ε, για την δέσμευση, τις αποθήκες δέσμευσης, σε ε, και αποθήκευσης. Ε. Δεν πρέπει να ενισχύσουμε τις παρουσές αποθήκες εφόσον μειώνεται, μειώνεται αντίστοιχε αποθήκες ε, στα δάση πώς η βιώσιμη χρήση των δασικών ε, πόρων θα έρθει στην πρώτη γραμμή και επίσης πώς θα μπορέσουμε να ε, σταματήσουμε την ε, απώλεια βιοπικιλότητας. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Έχετε περίπου 15 λεπτά για να απαντήσετε herra puheenjohtaja kiitoksia paljon hyvistä ja tiukoista kysymyksistä. Käyn lävitse. Ευχαριστώ πρόεδρε πολλές και δύσκολε οι ερωτήσεις. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όλα τα ερωτήματα. Να ξεκινήσω με τα δάση, διότι έγινε αναφορά. Το πιο σημαντικό εδώ είναι η βιωσιμότητα των δασών. Αυτό σημαίνει ορθή διαχείριση και όταν μιλάω για διαχείριση, εννοώ ότι θα πρέπει τα δάση να μπορούν να μεγαλώσουν. Το ξέρω αυτό και από τη δική μου εμπειρία, διότι είμαι ο ίδιος Γιώργος, έχοντας και σε εκτάσεις στην κατοχή μου, η οικογένειά μου δραστηριοποιείται σε δασικές περιοχές εδώ και 450 χρόνια. Και πάντα θεωρούσαμε ότι είναι σημαντικό να προστατεύσουμε το περιβάλλον μας έτσι ώστε η επόμενη γενιά να το βρει ακόμα καλύτερο από ό,τι εμείς. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για μας. Το δεύτερο έχει να κάνει με το θέμα της αποψήλωσης. Θα πρέπει να σταματήσουμε το φαινόμενο, να το περιορίσουμε. Υπάρχουν διάφορες ιδέες για το πώς μπορούμε να υποχρεώσουμε τους ε, εμπορικούς μας εταίρους να έχουν μια σωστή συμπεριφορά για το θέμα αυτό. Και σίγουρα θέλουμε αυτό στην Προεδρία μας να το τονίσουμε. Πώς μπορεί να γίνει αυτό. Η Φιλανδία πάντα πίστευε σε μια συνεργασία εμπορική που θα βασίζεται σε κανόνες είναι βασική αρχή μας. Είτε αφορά, αυτή, αυτό αφορά τα δάση, είτε την κυκλική οικονομία. Κάποιοι είπαν πώς μπορούμε να εγγυηθούμε την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας μας. Μέρος της βιομηχανίας μας ε, βασίζεται στη βιολογική οικονομία θα πρέπει να στραφεί προς νέες τεχνολογίες, να κάνει νέες επενδύσεις σε, σε νέους τομείς. Θα πρέπει δηλαδή και η βιομηχανία να παράγει προϊόντα με περιβαλλοντικός ορθό και φιλικό τρόπο. Και τα προϊόντα αυτά να μας βοηθήσουν να αντικαταστήσουμε στο μέλλον τα ορυκτά καύσιμα μεταξύ άλλων. Ε, είναι κάτι που πρέπει να γίνει στην Ευρώπη αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εξασφαλίσει ότι αυτό θα συμβεί και στα πλαίσια του διεθνούς εμπορίου. Το πολιτικό δημοσιονομικό πλαίσιο. Και εδώ ακούστηκαν πολλά ερωτήματα. Είναι σαφές ότι οι μεγάλες μας φιλοδοξίες ε, για τα ζητήματα τα περιβαλλοντικά και τα κλιματικά πρέπει να συνοδεύονται και από χρήματα, από χρηματοδότηση πάνε χέρι-χέρι αυτά. Γι' αυτό λοιπόν θέλουμε να συνεργαστούμε με την Κομισιόν, με τα κράτη-μέλη, έτσι ώστε να υπάρξει βεβαίως, μια ισότιμη συμμετοχή των κρατών μελών, δίκαιη, και να βεβαιωθούμε κυρίω ότι οι πυλώνες που έχουμε δημιουργήσει λειτουργούν, ε, εξυπηρετούν τους στόχους μας. Στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την μεταρρύθμιση τη κοινωνική πολιτική υπάρχουν πάρα πολλά θετικά στοιχεία που θα μας επιτρέψουν να πετύχουμε τους νέους στόχους μας, θα μας επιτρέψουν να απλοποιήσουμε μια σειρά από διαδικασίες και αυτό είναι σημαντικό για τη χώρα μας. Η απλοποίηση. Έχουμε νέες δυνατότητες ε, που μας προσφέρει η ψηφιοποίηση, στοιχεία που θα μας βοηθήσουν και στον τομέα των ελέγχων. θα δραστηριοποιηθούμε λοιπόν και στον τομέα αυτών. Ε, ο ρόλος της γεωργίας στο παγκόσμιο σύστημα είναι κεφαλαιώδης. Ε, το πιο σημαντικό εδώ είναι η διατροφική ασφάλεια. Πρέπει να υπάρχει βιώσιμη παραγωγή των τροφίμων για να μπορούμε να διατηρήσουμε τη βιοπικιλότητα και η διαδικασία αυτή πρέπει να είναι ισορροπημένη. Τι σημαίνει αυτό νέες τεχνολογίες γεωργικές να βασιστούμε στα πιο πρόσφατα στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα και τα στοιχεία αυτά, οι πρακτικές αυτές να αναπτύσσονται γρήγορα στην Ευρώπη. Έτσι μπορούμε να αυξήσουμε και την ανταγωνιστικότητά μας απέναντι σε άλλες οικονομικές ζώνες. Πολύ σημαντικό αυτό. Αυτό σχετίζεται και με το τι βεβαίως ε, καλλιεργούμε και πώς το καλλιεργούμε. Η άτυπη Υπουργική Σύνοδος Γεωργίας και Αλίας στο φθινόπωρο στο Ελσίνκι θα αφιερωθεί ακριβώς σε αυτό το θέμα. Πώς μπορούμε ε, ε, να δεσμεύσουμε, να αποθηκεύσουμε άνθρακα στο έδαφος Ταυτόχρονα βεβαίως ε, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την ανάπτυξη. Πρέπει αυτή η αποθήκευση να οδηγήσει σε περιβαλλοντικά και κλιματικά ωφέλη. Είναι πολυσχεδής η προσπάθεια, ε, αλλά πρέπει να την κάνουμε. Η δέσμευση λοιπόν του άνθρακα είναι πολύ σημαντική. Πρέπει να κάνουμε και περισσότερο στον τομέα της έρευνας γνωρίζουμε καλύτερα τι συμβαίνει ε, στο έδαφος από ότι στο υπέδαφος και, και πρέπει να βελτιωθεί, να βελτιωθούν οι γνώσεις μας εδώ. Έγινε αναφορά στις νήσους Όλαντ ε, και τι γίνεται ε, με τον Μπακαλιάρο εκεί. Βεβαίω, ε, σε ορισμένε περιοχέ υπάρχει επιδείνωση κατάσταση, αλλά όχι παντού. Ε, το συζητούμε αυτό με την Κομισιόν. Ε, χρειάζονται οι απαραίτητε επιστημονικέ πληροφορίε, τα στοιχεία για το τι γίνεται με τα διάφορα αλλιευτικά είδη, τα διάφορα ψάρια. Υπάρχουν πολλές διαφορές μεγάλες από περιοχή σε περιοχή. Στον τομέα της αλίας, όπως είπα, οι επιστημονικές νοματεύσεις ε, θα, είναι η βάση της δράσης μας. Θέλουμε βιώσιμη αλία, θέλουμε βιώσιμα αλλιευτικά αποθέματα και πρέπει πάντα να βλέπουμε πιο μακριά στον χρόνο. Και εδώ βεβαίως η Κομισιόν έχει πολλές αρμοδιότητες. Τώρα, για το Μερκοσούρ. Βεβαίως ε, αυτή η συμφωνία δημιουργεί πολλές προκλήσεις. Λίγες μέρες πριν ε, το Συμβούλιο Αλίας και Γεωργίας λάβαμε αυτό το έγγραφο και βεβαίως ε, τα κράτη-μέλη θα το αξιολογήσουν, θα το αξιολογήσουν το καθένα την πλευρά του, ε, κατά πόσο δηλαδή αυτή η συμφωνία θα επηρεάσει και με ποιον τρόπο τη γεωργία. Αυτό θα πάρει χρόνο, αυτή η αξιολόγηση. Βεβαίως υπάρχουν πολλά ερωτηματικά, προφανώς. Θα πρέπει να απαντηθούν τα ερωτηματικά αυτά και αυτό είναι βέβαιο. Και βέβαια θέλουμε να συνεργαστούμε και με την Κομισιόν και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ιδιαίτερα με την Κομισιόν η οποία έχει σημαντικές εξουσίες εδώ, Θέλουμε λοιπόν, λοιπόν να μελετήσουμε όλα αυτά τα ζητήματα πολύ προσεκτικά και μετά από ε, εξαιρετικά προσεκτικές διαπραγματεύσεις θα φτάσουμε και σε αποφάσεις. Αντιλαμβάνομαι βεβαίως τις ανησυχίες σας, τις καταλαβαίνω πολύ καλά. Θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει σεβαστή η Συμφωνία των Παρισίων. Θα πρέπει πάντα να έχουμε κατά νου αυτή τη συμφωνία. Υπήρξε και ένα ερώτημα για τα ζανιοκτώνα. είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι μια ακρογωνία λήθος ε, της ε, μεταρρύθμισης της κοινωνικής πολιτικής, ένας ακρογωνίας λήθος, είναι η βιοπικιλότητα. Και αυτό έχει να κάνει με όλες τις πτυχές. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη μας και τα έντομα και βεβαίω εδώ μπαίνει το θέμα τη επικονίαση, όπω αντιλαμβάνεστε. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να προστατεύσουν τη βιοπικιλότητα σε διάφορα κράτη-μέλη. Είναι μια δουλειά, μια προσπάθεια να εξελίξει. Τώρα, η πράσινη αρχιτεκτονική. Αυτό είναι ένα θέμα που συνδέεται με τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ είχαμε ήδη μια μακρά συζήτηση, μια καλή συζήτηση για το θέμα αυτό στην πρώτη, στο πρώτο Συμβούλιο Γεωργίας και Αλίας. Μας δίνει τη δυνατότητα να προβούμε στις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις και ταυτόχρονα να δώσουμε ευελιξία στα κράτη-μέλη. Τα κράτη-μέλη δηλαδή να λάβουν υπόψη τους τις όποιες, ε, όποιους φυσικούς περιορισμούς, τις ιδιαιτερότητες που υπάρχουν σε διάφορες χώρες οι οποίες είναι αναπόδραστες. Είναι σωστή η προσέγγιση πάντως ε, εδώ. Να δώσω ένα παράδειγμα. Στη Φιλανδία, και το λέω και ως Γιωργός αυτό, στα πλαίσια του δεύτερου πυλώνα, στη Φιλανδία, έχουμε εισαγάγει πολύ σημαντικά κίνητρα και έτσι 90% των γεωργών έχουν αποφασίσει να ακολουθήσουν αυτές τις λύσεις. Όταν προσεγγίζουμε την κατάσταση σε μια χώρα πρέπει να βρίσκουμε εστιασμένες λύσεις για να επιτευχθεί ο στόχος. Να λάβουμε υπόψη μας δηλαδή τις τοπικές συνθήκες, τις τοπικές προκλήσεις κάθε φορά. Αυτό είναι κάτι που δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Και να πω και δύο λόγια για τα ζυζανιοκτώνα και τη διαδικασία αδειοδότησης. Η ΕΦΣΑ είναι η αρμόδια αρχή, ε, η οποία πρέπει να χρηματοδοτηθεί περαιτέρω. Ε, κάνει πολύ σημαντική δουλειά η ΕΦΣΑ, αποτελεί τη βάση ε, για την διαχείριση κινδύνου και τις αποφάσεις που παίρνουμε και ως Προεδρία θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι η ΕΦΣΑ θα έχει ό,τι χρειάζεται για να κάνει τη δουλειά της. Διότι είναι πολύ σημαντικό το επιστημονικό της έργο. Ευχαριστώ πολύ. Thank Ευχαριστώ πολύ. Τώρα μπαίνουμε στο δεύτερο γύρο ερωτήσεων. Αυτός ε, θα χωριστεί σε δύο τμήματα. 13 βουλευτές, πρώτα 7 και μετά ε, θα απαντήσει ο κύριος Υπουργό και μετά οι άλλοι έξι, γιατί διαφορετικά θα έχετε πάρα πολλές ε, ερωτήσεις και θα είχατε και ένα καλό πρόσχημα για να μην τις απαντήσετε. Γι' αυτό λοιπόν αποφασίσαμε ότι καλύτερα θα ήταν να μοιράσουμε στα δύο τις ερωτήσεις. Αλεξάνδρου Μπενχούμπερ από το ΕΛΚΑ. Αξιότιμε Πρόεδρε, αξιότιμη Υπουργέ, σα ευχαριστώ πολύ για την εισαγωγή σα παρέμβαση και την παρουσίαση ενό φιλόδοξου προγράμματο. Είστε άλλωστε από ένα κόμμα με περιβαλλοντικέ ανησυχίε, είστε αγρότης και εσεί μιλήσατε για την προστασία τη βιοπικιλότητας και τη βιωσιμότητα. Σε ό,τι αφορά τη βιοπικιλότητα θέλω να πω ότι είναι πολύ σημαντική η οδηγία για την ε, Φλωρίδα και Πανίδα που δεν έχει τροποποιηθεί μετά τη δεκαετία του 90. Υπάρχουν όμως σημαντικά προβλήματα. Θέλουμε να υπάρχει καλή συμβίωση ε, του ανθρώπου, του περιβάλλοντος, ε, της λόγιδας και Πανίδας. Ε, όμως Υπάρχουν αυτά τα οικοσυστήματα τα οποία προστατεύονται με αυτή την οδηγία, αλλά υπάρχουν ε, ε, επιπτώσεις λόγω της αύξησης του πληθυσμού ε, και με, τη, με τους ποταμούς. Υπάρχει πρόβλημα στη βιοπικιλότητα, χλωρίδα, πανίδα. Έχουμε το πρόβλημα επίσης με την αύξηση του πληθυσμού των λύκων στην Ευρώπη που καταπατούν ε, περιοχές, ιδίως ε, στις ε, ορεινές περιοχές και όπου πραγματικά δεν υπήρχε παρουσία τους. Έχουν 17.000 παραδείγματος χάρη τέτοιους, τέτοια ζώα. Τι έχετε να μας πείτε για όλα αυτά. Ευχαριστώ. Αλλά παρακαλώ να μην υπερβαίνετε το ένα λεπτό για τις ερωτήσεις σας. Σίλντα, σοσιαλιστές και δημοκράτες. Αξιότιμη κύριε Υπουργέ, Είμαστε οι πρώτοι που απαγορεύσαμε τη γλυφοζάτη από το 2020. Υπάρχουν ε, καλοί βάσιμοι λόγοι ε, και υπήρξε και ε, συμφωνία και εκ μέρους της κοινή γνώμης σε ό,τι αφορά αυτό. Τι άλλα μέτρα θα μπορούσαν να ληφθούν σε ό,τι αφορά τη χρήση αυτών των τοξικών προϊόντων και τι υποκατάστατα, τι λογικές συναλλακτικές θα μπορούσαν να βρεθούν που είναι θετικές για το περιβάλλον αλλά και για τους καταναλωτές. Εσείς θα καταθέσετε τέτοιες πρωτοβουλίες ό,τι αφορά την έρευνα και την ανάπτυξη τέτοιων εναλλακτικών για να αντικατασταθούν αυτά τα χρησιμοποιούμενα μέχρι τώρα φυτοφάρμακα και ζυζανιοκτών. Ευχαριστώ. Renew Martin Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμε Υπουργέ. Η κοινωνική πολιτική αφορά το κλίμα, αφορά τη βιοπικιλότητα, τα χημικά, αλλά και την καλή μεταχείριση των ζώων. Μίλησαν κάποιοι για την για δέσμευση του άνθρακα και δεν θα επανέλθω, αλλά θα μιλήσω για κάτι που προέρχεται, που συνδέεται με τον άνθρακα και τα θερμοκηπιακά αέρια. Πώς επηρεάζονται τα ζώα. Τι θα κάνετε εσείς ως Προεδρία στο πλαίσιο τη μεταρρύθμιση τη και πολιτικής, πολιτική, ιδίω ε, έχοντα υπόψη και την αποψήλωση του Αμαζονίου των δασών. Τι θα κάνετε λοιπόν σε σχέση με την καλή μεταχείριση των ζώων και την ε, εντατική κτηνοτροφία. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα δάση, με κανοποίησαν αυτά που είπατε για τη βιώσιμη αηφόρο δασοκομεία. Υπάρχει όμως μια σημαντική πρόκληση και σε τρίτες χώρες αλλά και εντός Ένωσης λόγω της αποψήλωσης. Το βλέπουμε και στη δική μας τη χώρα, σε περιοχές που ανήκουν και στο δίκτυο Natura 2000. Θα μπορούσατε να κάνετε κάτι στον Προεδρία, για να πιέσετε προς ε, καλύτερη επιβολή για εφαρμογή και, επιτρο... Ε, και προστασία των ε, εδαφών Natura. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Πολλές ε, ερωτήσεις έγιναν για την κοινή γεωργική πολιτική ήδη και για μια κοινή προσέγγιση που θα μπορούσαμε να βρούμε. Σίγουρα η προστασία της βιοπικιλότητας θα είναι δυνατή αν υπάρχει μια κοινή προσέγγιση σε ό,τι αφορά ε, την ε, γεωργία. Θα ήθελα λοιπόν να μας πείτε συγκεκριμένα τι θα κάνετε για την ε, ε, διάσκεψη της Κίνας ε, στα τέλη του έτους ε, και τη συμφωνία που θα συζητηθεί εκεί, τι θα προτείνετε και πώς μπορεί να εξασφαλιστεί ο γετικός ρόλος, ο πρωτοποριακός ρόλος της Ένωσης, ότι αυτή η προστασία της βιοποικιλότητας, ότι δεν αφορά τη συμφωνία ε, Μερκοσούρ για την προστασία, ε, την τη φυτοπροστασία, τι μέτρα θα μπορούσαν να, να βελτιώσουν την κατάσταση, αλλά να εξασφαλίσουν και την προστασία των καταναλωτών Πώ πώς θα εξασφαλίσουμε τα πρότυπα ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τι έλεγχοι και τι εξασφαλίσεις μπορούμε να έχουμε. Σεζάρ Λουενά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε, κύριε Υπουργέ, αναφερθήκατε στη, στο ΠΙΔΕΛΤΑΠΗ. Ε, εδώ βρισκόμαι. Νομίζω ότι η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τα εκεί πηγαίνει, δηλαδή προς την απλούστευση, την ευελιξία. Ωραία όλα αυτά, αλλά εγώ θα ήθελα όμως να μου πείτε ότι ενώπιον του Συμβουλίου θα υπεραμεινθείτε της μη περικοπής των κονδυλίων της ΚΑΠ. όσον αφορά τη δασοπονία, δασοκομεία, μπορείτε να μας αναφέρετε πιο συγκεκριμένα μέτρα για την ανάπτυξη της συμβολής της γεωργίας, της δασοπονίας και της καταπολέμησης κλιματικής αλλαγής σε σχέση και με κάτι άλλο που είπατε και εσείς, την ανάπτυξη της βιοοικονομίας. Επίσης, για το Μερκοσούρ, ε, οι προστατευόμενες, ε, οι ονομασίες προέλευσης προστατεύονται. Ναι, θέλουμε να εξακολουθήσει η προστασία αυτή ε, και αυτό που είπα προηγουμένως, οι πόροι της ΚΑΠ να μην πειραχτούν από το Συμβούλιο. Ευχαριστώ πολύ Μάρτιν για τους πράσινους. Κύριε Υπουργέ, μιλήσατε για την τη Πολιτική. Ε, και δίνουμε ε, πληρωμές ε, στρεματικές ενισχύσεις ε, οι οποίες ανέρχονται στα δύο τρίτα των γεωργικών κονδύλων. Τι κάνουμε για το κλίμα, τι κάνουμε για το περιβάλλον. Δεν είναι νομίζω η μεταρρύθμιση όπως παρουσιάζεται αρκετά φιλόδοξη και πραγματικά θα πρέπει να κάνουμε τελείως διαφορετικά πράγματα κατά της απώλειας της βιοπικιλότητας μέσα και για τον να έχουμε περικοπές τάξης 30% και εσείς στη Φιλανδία ωφελείστε περισσότερο, αλλά νομίζω ότι χρειαζόμαστε για το δεύτερο πυλώνα περισσότερα χρήματα, χρειαζόμαστε για την οικολογική γεωργία περισσότερα χρήματα, όταν θα αρχίσει να ισχύει από το χρόνο και ο νέος κανονισμός. Επίσης ε, για την αντοχή στα αντιβιωτικά, ε, ξέρουμε ότι αναπτύσσονται συνέχεια νέα αντιβιωτικά Έχουμε εισαγωγές ε, υλικών ε, που είναι προϊόντα γενετικής μηχανικής. Ε, τι κάνει το Συμβούλιο Κομισιόν με την εισαγωγή τέτοιων προϊόντων. Ευχαριστώ. Μαρία Σπυράκη από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε κύριε Υπουργέ. Θα ήθελα να επιμείνω σε κάποια θέματα, τα οποία ήδη αναφέρθηκαν βέβαια, που όμως πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουμε περαιτέρω πληροφορίες από αυτόν. Η χρηματοδότηση πρώτα απ' όλα. Φυσικά, στα πλαίσια της αντιμετώπισης των κλιματικών στόχων. Νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε το ενδεχόμενο επιπρόσθετης ε, χρηματοδότησης ε, της ε, ΚΑΠ. Έγινε μια αναφορά σε ένα δις για τη γεωργική οικονομία που θα δοθούν στους ενίδη δανείων. Αλλά πόσοι θα είναι και ποιοι θα είναι αυτοί οι γεωργοί. Εγώ πρέπει να σας πω ότι μονάχα 7% των ε, γεωργών καταφέρνουν να ζουν πραγματικά από την ε, δουλειά τους. Ε, τι... Ε, και μόνο αυτοί είναι που μπορούν να αποκτήσουν επιπλέον δεξιότητες μέσα από τα σχετικά προγράμματα. Τι θα κάνετε έτσι ώστε να, αρχίσει, ε, να αρχίσουν να εφαρμόζονται όλα αυτά τα προγράμματα στα κράτη-μέλη. Ευχαριστούμε πολύ για αυτό το πρώτο γύρο ερωτήσεων. Δέκα λεπτά έχετε για να απαντήσετε. Κοίταξε, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για τις εξαιρετικές ερωτήσεις. Όλο και με δυσκολεύετε. Λοιπόν, κάποιες ερωτήσεις εμπίπτουν στο χαρτοφυλάκιο άλλων ε, υπουργών, όπως αυτή η οδηγία για τα οικοσυστήματα. Γιατί είναι αρμοδιότητα του Υπουργού περιβάλλοντος και θα είναι αυτός φαντάζομαι που θα σας απαντήσει καλύτερα για αυτό το θέμα. Σίγουρα υπάρχουν αλλαγές στο περιβάλλον, το ζωικό κεφάλαιο αλλάζει, αλλάζουν διάφορα, διάφορες συνθήκες και καταστάσεις και όλα αυτά πρέπει να τα λάβουμε υπόψη. και για τις περιοχές του Natura 2000 ε, είναι αρμοδιότητα ε, του Υπουργού Περιβάλλοντος. Στη Φιλανδία ε, και εμείς πρέπει να εφαρμόσουμε τις υποσχέσεις που δώσαμε και τις δεσμεύσεις που πήραμε τις κάνουμε πράξη και αυτό θα κάνουμε. Είναι πράγματι πολύ σημαντικό για την Προεδρία μας ότι αυτή τη γλυφοζάτη Συμφωνώ και εγώ ότι χρειαζόμαστε εναλλακτικά ζυζανιοκτώνα φυτοφάρμακα και πρέπει να αναπτυχθούν νέα ασφαλή ε, φυτοφάρμακα και νέες τεχνολογίες να προωθηθούν. Να δούμε κατά πόσο χρειάζονται, πού χρειάζονται και πού δεν χρειάζονται ε, αυτά τα ζυζανιοκτώνα στην κυρία και είμαι ανοιχτός να το συζητήσουμε πολύ σοβαρά το θέμα και για την κυβοζάτη και για τα ε, φυτοφάρμακα τα υπόλοιπα. Ε, το θέμα δεν είναι μόνο η χρήση τους, ότι τα χρησιμοποιούμε, αλλά και το πώς, με ποιο τρόπο τα χρησιμοποιούμε. Σίγουρα υπάρχουν διαφορετικές τεχνικές, διαφορετικές τεχνολογίες και όλα αυτά ε, επηρεάζουν με διαφορετικό τρόπο το περιβάλλον. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά. Η καλή μεταχείριση των στον κάτι που αναφέρθηκε από αρκετού βουλευτέ. Είναι ένα μείζον ζήτημα. Τι μιλάμε για Μερκοσούρ, εξαγωγές των ζώων, κτηνοτροφία, πάχνηση και οτιδήποτε. Το σημείο κίνηση πάντα είναι η καλή μεταχείριση των ζώων και θα αναλάβουμε δράση στο μέτωπο αυτό. Πάκτα sunt servanta. Αυτό πρέπει να κάνουμε και θα το κάνουμε. Επανέρχομαι στο Μερκοσούρ. Υπάρχουν ρήτρες ε, διασφάλισης που πρέπει να τηρηθούν. Παραδείγματο χάσω ό,τι αφορά την ε, μικροβιακή αντοχή, υπάρχει μια τέτοια ρήτρα. Γιατί υπήρξαν ερωτήσεις σε σχέση με τα σχετικά αντιβιωτικά. Ε, εγώ δεν είμαι υπέρ της προληπτικής χρήσης αντιβιωτικών τα αντιμικροβιακά ή τα αντιβιωτικά χρησιμοποιούνται όχι για πρόληψη αλλά για θεραπεία νόσων. Πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε και εδώ ε, να προστατεύσουμε την υγεία των ζώων. Αλλιώς θα φτάσουμε σε μια κατάσταση που δεν θα έχουν πλέον καμία ε, επίδραση οι ουσίες αυτές. Θα έχουν χάσει τη δράση τους. Πάντως το θέμα αυτό γενικά είναι πάρα πολύ σημαντικό και χαίρομαι που ετέθη. Οι καταναλωτές τώρα. Βεβαίως και θέλουν να γνωρίζουν τις διαδικασίες, τις διεργασίες ε, παρασκευής των ε, τροφίμων, τι συστατικά περιλαμβάνουν, φυσικά και η ε, αντοχή στα αντιμικροβιακά είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. κοινή γεωκή πολιτική, φιλοδοξίες, ε, ιδίω στα περιβαλλοντικά ζητήματα. Υπάρχουν φιλοδοξία. Θέλουμε να προωθήσουμε τη μεταρρύθμιση τη κοινής πολιτική πολιτικής και θα παραμείνουμε φιλόδοξοι. Όταν αυξάνεται βέβαια ε, τα επίπεδα φιλοδοξίας, δεν θα πρέπει να μειώνονται τα επίπεδα της χρηματοδότησης. Αυτά πρέπει να συμβαδίζουν φιλοδοξία με χρηματοδότηση. Πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία. Το έχω πει ήδη τρεις φορές. Και το έχει πει και η Προεδρία κατά το παρελθόν, το λέω και εγώ ακόμη μια φορά. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώ ε, ποιος βουλευτής ε, το είπε, αλλά κάποιος μίλησε για την ε, χρηματοδότηση της ξένης γεωργικής πολιτικής και μου ζήτησε να διασφαλίσω την επαρκή χρηματοδότηση. Σας το υπόσχομαι. Θα φροντίσω να υπάρχει επαρκής χρηματοδότηση για την κοινή γεωργική πολιτική. Το έχει πει και δηλώσει η Φιλανδική Προεδρία ότι αυτό είναι προτεραιότητα. Σίγουρα πρέπει να υπάρχουν διαφοροποιημένα εργαλεία χρηματοδοτικά για να προσεγγίσουν όλους τους αγρότες και να αντιμετωπίσουν ε, τις διαφορετικές συνθήκες. Είναι καλό να υπάρχει ποικιλία, να υπάρχουν περισσότερες στις μιας μορφές χρηματοδότησης Και ξέρετε, εγώ για να βάλω τώρα, να σας μιλήσω από την ιδιότητα του αγρότη, και γιατί κοιτάζομαι και στον καθρέφτη και βλέπω έναν αγρότη μπροστά μου, πρέπει σίγουρα να αναπτύξουμε δεξιότητες ή να βελτιώσουμε τις δεξιότητες. Δεν μπορούμε να σαλιώνουμε το δάχτυλό μας για να δούμε προς τα που φυσάει ο αέρας. Πρέπει να βελτιώσουμε τις δεξιότητές μας. Και Χαίρομαι ιδιαίτερα που έγινε λόγος για τους ε, νέους αγρότες και την ε, ανάπτυξη τον Είναι, Γεωργία, κάτι που μου είναι ιδιαίτερα προσφυλές. Και πρέπει να κάνουμε τους αγρότες να συνεχίσουν να πιστεύουν στο μέλλον και ιδίως τους νέους αγρότες για να συνεχίσουν να παράγουν τρόφιμα για εμάς ε, στο μέλλον και να είναι ασφαλή αυτά τα τρόφιμα. Η έρευνα λοιπόν και η επένδυση ε, στην έρευνα και στην άπτυξη είναι σίγουρα κάτι πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ για την παρουσία σας. Πρέπει να σας πω ότι ανησυχώ λίγο με αυτά που λέτε. Λέτε ότι θα είστε ε, έξι μήνες ε, ε, επικεφαλής του Συμβουλίου. Αυτό μας ευχαριστεί, αλλά μετά ακούω διάφορα πράγματα για την ΚΑΠ και λίγο προβληματίζομαι. Μου λέτε ότι όλοι οι υπουργοί υπεραμείνονται του, ε, τον προπολογισμό, αλλά εμείς έχουμε 15% στην πρόταση που ε, μας ε, φέρνετε 15% μείον για την γεωργία, 7% μείον για τη συνοχή ε, και επομένως από ό,τι καταλαβαίνω ότι θα έρθετε και εσείς μαζί μας αυτόν τον αγώνα που δίνουμε για την, την επιπλέον χρηματοδότηση. Επίσης, Λέτε ότι όσον αφορά ε, την στρατηγική όλα πάνε καλά, αλλά εγώ αντιθέτως έχω την εντύπωση ότι εδώ και δέκα μήνες ε, στην ουσία κάνουμε σημειωτών ε, και δεν σαν καθόλου υπόψη οι προτάσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Νομίζω ότι όσον αφορά τη βιοπικιλότητα, όσον αφορά την ανθρώπινη υγεία, την ασφάλεια, την διατροφική, το περιβάλλον, όσον αφορά το συνολικό περιβαλλοντικό, ε, περιβαλλοντικό σχήμα δεν ε, είμαστε στο ύψος των καταστάσεων με την νέα ΚΑΠ. Θα πρέπει ίσως να ξαναδούμε το μοντέλο της ε, ΚΑΠ και πραγματικά αυτά τα οποία λαμβάνουν χώρα τώρα και οι προτάσεις που βλέπουμε δεν είναι στο ύψος των φιλοδοξιών που θα πρέπει να έχει η Γεωργία. Η Μαρία Σοράροβα όμως, που είσαι Μαρία. Καλώς ορίσατε κύριε Υπουργέ για την ε, ΚΑΠ και εγώ πολύ σύντομα. Είναι γεγονό ότι είναι φιλόδοξη η μεταρρύθμιση ε, και οπωσδήποτε θέλουμε ε, να ενσωματωθούν εδώ και οι αποφάσεις του θεματολογίου του 2030 καθώς επίσης και τη Συμφωνία των Παρισίων. Εγώ θα ήθελα να σας πω ότι ανησυχώ όσον αφορά την ευελιξία των εθνικών στρατηγικών ε, σχεδίων και κατά πόσον αυτά, αυτή μπορεί να οδηγήσει σε εν μέρει επανεθνικοποίηση των ε, πολιτικών. Και όσον αφορά τις ε, κοινές, ε, τα κοινά πρότυπα, θα πρέπει να υπάρχουν τέτοια κοινό πρότυπα και στις, ε, στα εθνικά προγραμματικά σχέδια. Επίσης, εκτός από την eco-conditionality, θα πρέπει να υπάρξουν και κάποια κίνητρα, κάποια μέτρα κινητροδότησης για αυτούς τους γεωργούς που θέλουν να κάνουν περισσότερο. Ε, μήπως τα eco-schemes θα πρέπει να γίνουν υποχρεωτικά. Επίσης, δεν πιστεύετε ότι θα πρέπει οπωσδήποτε και στις υπόλοιπες πολιτικές να ληφθεί υπόψη και η ισότητα των φύλων έτσι ώστε ε, και οι γυναίκες να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες με τους άντρες. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ορελιά Μπενιέ για την ομάδα ID. Κύριε Υπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι, η το πρόγραμμα της Φιλανδικής Προεδρίας μας προβληματίζει σχετικά με το τι θα ακολουθήσει. Μας λένε ότι ο προστατευτισμός δημιουργεί πρόβλημα στην ευρωπαϊκή οικονομία. Ωστόσο όμως ε, οι πολίτες της Ευρώπης ζητούν κάτι αντίθετο. Ζητούν περισσότερα τοπικά προϊόντα και μεγαλύτερη χνηλασιμότητα. Ξέρουμε ότι ε, ε, έχουν μπει στην ευρωπαϊκή αγορά από τον Καναδά πολλά προϊόντα προϊόντα τα οποία περιλαμβάνουν στοιχεία τα οποία εδώ και πάρα πολύ καιρό έχουν ή σε την ε, Ευρώπη. Επίσης χρησιμοποιούν, ε, χρησιμοποιούνται στην ε, Φιλανδία πρέπει να πω κάποιες ουσίες οι οποίες έχουν απαγορευτεί όσον αφορά την εντατική γεωργία. Δεν είναι δυνατόν να επιτρέψουμε να μην χρησιμοποιούν οι γεωργοί μας προϊόντα τα οποία και ουσίες που δεν έχει αποδειχθεί η επικίνδυνοτητά τους. Αυτά θα πρέπει να τα αντιμετωπίσετε ως Προεδρία. Ευχαριστώ. Αντρέα Ζεκάμπ Γκουε. Ευχαριστώ πολύ κύριε ε, Υπουργέ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και να σας συγχαρώ γιατί την προηγούμενη εβδομάδα ε, στην, στο Συμβούλιο Γεωργίας ξεκινήσατε τη συζήτηση όσον αφορά τον ε, χρόνο μεταφοράς των ζώων και τη μεταφορά των ζώων στη διάρκεια του καλοκαιριού γιατί έχουμε δει περιπτώσεις όπου ζώα πηγαίνουν από το ένα μέρος στο άλλο υπό 40 βαθμούς υποσκιά καθώς επίσης ε, ε, ξέρουμε την περίπτωση αυτών των πολλών χιλιάδων αρνιών που με απίστευτα κακές συνθήκες ακόμα ε, δεν έχουν φτάσει στο Κουβέιτ. Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να μου πείτε με ποιο τρόπο θα καταβάλλετε προσπάθειες έτσι ώστε να σταματήσουν αυτές οι τόσο κακές μεταφορές ε, και με ποιο τρόπο θα αντιμετωπίσετε τις αντιστάσεις ε, του ομολόγου σας Ρουμάνου Υπουργού Γεωργίας. Θα δώσουμε τώρα το λόγο στην κυρία Ντανούτσκα ε, για το ECR στο δεύτερο γύρο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, ήθελα να είμαι εξαιρετικά πειθαρχημένη και να μην ξεπεράσω το χρόνο. Γι' αυτό το ξέχασα ένα ερώτημα προηγουμένως και θα το θέσω τώρα. Όταν μιλάμε για τα δάση και την νόσιμη ενέργεια, την προστασία του περιβάλλοντος, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι θα πρέπει να προλάβουμε καταστάσεις όπου καταστάσεις που υπαρκτές, έτσι, υπαρκτές σε κάποια μεγάλα κράτη-μέλη, όπου υπάρχει αποψήλωση μεγάλης κλίμακας. Μόνο και μόνο γιατί, για να δημιουργήσουμε αιωλικούς, ε, αιωλικές εγκαταστάσεις. Αυτό πραγματικά είναι παράλογο. Δεν μπορεί να μην μπορούμε να τις βάλουμε αλλού αυτές τις αιωλικές εγκαταστάσεις, τα αιωλικά πάρκα, χωρίς να καταστρέφουμε δάση. Λοιπόν, όταν θα συζητήσουμε τη δασοκομεία, ε, και την προστασία των δασών και πώς θα επιτευχθεί ο στόχος ε, των μηδενικών εκπομπών, καλό είναι να έχουμε κατά νου και αυτές τις περιπτώσεις. Ευχαριστώ. Τελευταίο ερώτημα. Ελεονόρα Ευή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε κύριε Υπουργέ. Μιλήσατε προηγουμένως στη, για το θέμα της μικροβιακής αντίστασης. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο πλέον έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις. 33.000 ε, και παραπάνω είναι τα άτομα που χάνουν τη ζωή τους από το πρόβλημα αυτό κάθε χρόνο στην Ευρώπη και το 2050 θα έχουν φτάσει στα 10 εκατομμύρια από ό,τι λένε διάφορες μελέτες. Ε, και το, ε, το φαινόμενο αυτό ακριβώς προέρχεται ε, και από την απαράλογη χρήση των αντιβιωτικών καθώς επίσης και την εντατική κτηνοτροφία που εν τέλει οφείλεται και για την μείωση της βιοπικιλότητας στην, στο, στην Ευρώπη είναι πάνω από 300.000 τα ζώα τα οποία βρίσκονται σε εχμαλωσία. Ένα εκατομμύριο 200.000 υπογραφές έχουν μαζευτεί ε, όσον αφορά το θέμα αυτό. Θα ακούσετε εσείς τους ανθρώπους αυτούς που έχουν υπογράψει τέτοιου είδους ε, ε, καταδικαστικές για την γεωργία, την εντατική γεωργία αποφάσεις και κείμενα. Πώς θα αντιμετωπίσετε τέτοιου είδους κείμενα εσείς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δέκα λεπτά για να απαντήσετε κύριε Υπουργέ. που puheenjohtaja, kiitos jälleen kysymyksistä. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ ακόμα μια φορά για τις ερωτήσεις σας. Θα προσπαθήσω να απαντήσω με τη σειρά λίγο πολύ για τη χρηματοδότηση βεβαίως υπάρχουν πολλά ερωτηματικά. Ε, αυτό είναι λογικό και είναι και καλό. Είναι κρίσιμο το ζήτημα που αντιλαμβάνεστε για το μέλλον της πολιτικής μας. Η συνοχή είναι κρίσιμη για μας. Να σας πω ότι η χρηματοδότηση παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στον τομέα τη κοινή πολιτική ε, και συζητείται σε επίπεδο Υπουργών Γεωργία, αλλά οι αποφάσει θα παρθούν σε επίπεδο αρχικών κρατών και κυβερνήσεων. Οι φιλόδοξοι περιβαλλοντικοί στόχοι πάντω ε, μπορούν να επιτευχθούν μόνο με την ανάλογη χρηματοδότηση. Έχουν προταθεί κάποιε περικοπέ ε, στο δεύτερο πυλώνα και αυτό δημιουργεί δυσκολίες. Πρέπει να υπάρξει οπωσδήποτε ισορροπία μεταξύ των φιλοδοξιών που έχουμε θέσει ε, και της χρηματοδότησης για να επιτευχθούν οι στόχοι μας. Βεβαίως και ε, χρειάζεται βιώσιμη ανάπτυξη, χρειάζεται ταυτόχρονα ε, και ένα εισόδημα αξιοπρεπές για τους γεωργούς πρέπει πολλά να γίνουν και στον τομέα της διαχείρισης. Εκεί χρειάζεται απλότητα και ευελιξία. Εμείς ε, θέλουμε να έχουμε φιλόδοξους στόχους και βεβαίως πρέπει να, υπάρχει, να υπάρχουν προϋποθέσεις για τις όποιες ενισχύσεις με περιβαλλοντικές απαιτήσεις. Ναι στην ευελιξία λοιπόν, αλλά με κλιματικές δράσεις, κλιματικές δράσεις εστιασμένες ανάλογα με τις χώρες. Χωρίς επανεθνικοποίηση της πολιτικής μας βέβαια. Έχουμε κοινούς κανόνες, έχουμε κοινούς στόχους, αλλά πρέπει να βρούμε έξυπνους τρόπους εφαρμογής αναχώρα. Σε ό,τι αφορά την ευημερία των ζώων και τα, τις μεταφορές ε, μεγάλων αποστάσεων. Βεβαίως και είναι σοβαρό το θέμα. Εγώ το παίρνω πολύ στα σοβαρά, όπως είπα και στην αρχική μου ομιλία, αυτά τα κενά, αυτές οι ελλείψεις που έχουν διαπιστωθεί ε, δεν είναι αντάξια της εποχής στην οποία ζούμε. Πρέπει ο καταναλωτής να γνωρίζει ότι οι προϋποθέσεις Καθόλου την αλυσίδα παραγωγής και διανομής είναι κατάλληλες και οι προδιαγραφές γίνονται σεβαστές. Εμείς παρακολουθούμε την κατάσταση για τη συγκεκριμένη υπόθεση ως Προεδρία και θα συζητηθούν περαιτέρω τα ζητήματα αυτά στη συνεδρία των κτηνιάτρων των επικεφαλής κτηνιατρικών υπηρεσιών. Η διατροφή η ευρωπαϊκή είναι υψηλής ποιότητας. και βεβαίω ε, παρακολουθούμε στενά τις αγωγές από τρίτε χώρες, η αρχή της προφύλαξης, ε, η δημόσια υγεία ε, είναι κριτήρια τα οποία μας οδηγούν συχνά να αποσύρουμε τέτοια προϊόντα από την αγορά. Αυτό να μην το ξεχνάμε. Έτσι πρέπει να αντιδρούμε και να επανέλθω στο θέμα της αποψήλωσης. Ε, λέχθη σωστά νωρίτερα ότι συχνά τα δάση είναι θύματα της ε, ε, κατασκευαστικής ε, βιομηχανίας. Πρέπει εμείς όμως να δώσουμε έμφαση στην αναδάσωση. Έχουμε παράδοση στη Φιλανδία εμείς. Όταν χρησιμοποιείται ένα δάσος για οποιοδήποτε σκοπό, πρέπει στη συνέχεια να αναζωογονωθεί αυτή η περιοχή με νέο δάσος ή κάποια άλλη περιοχή αντίστοιχη. Αυτή είναι η αρχή ε, που μεταφράζεται και σε νόμο στη χώρα μας. Είναι και ένας τρόπος ε, να βελτιωθεί η ανάπτυξη των δασών. Και τέλος, Εμείς ε, δεν επιτρέπουμε κάποιες συγκεκριμένε ε, μορφές εντατικής ε, κτηνοτροφίας στην Ευρώπη, με τα πουλερικά παραδείγματος χάρη και τις, τα μικρά κλουβιά. Ε, πρέπει πάντα να βρίσκουμε τρόπους για να βελτιώνεται η κατάσταση, προϋποθέσεις, συνθήκες ευημερίας των ζώων και βεβαίως όλα αυτά λαμβάνοντας υπόψη για τη διατροφική ασφάλεια και πρέπει βεβαίως ε, τα προϊόντα που εισάγουμε από άλλες χώρες εκτός Ευρώπης ε, να πληρούν παρεμφαρείς προϋποθέσεις με τις δικές μας. Δύσκολο ζήτημα. Αλλά είναι ευθύνη που μας βαραίνει όλους. Ευχαριστώ πολύ. Ε, αν δεν έχω κάνει δεν απαντήσατε σε μια ερώτηση σχετικά με τη Συμφωνία για τη Βιοποικιλότητα στην Κίνα. Ερώτηση που έθεσε η κυρία Σνάιντερ. Εκτός και αν θα την απαντήσει ο συνάδελφός σας που είναι υπεύθυνο για το περιβάλλον. Ωραία, θα την κρατήσουμε λοιπόν την ερώτηση για αύριο. Α, μπορώ να προσθέσω κάτι, ναι, φυσικά. Κύριε Πρόεδρε, πράγματι Πρόκειται για ένα ερώτημα το οποίο αφορά τον ε, ε, Υπουργό Εξωτερικών και τον Υπουργό Περιβάλλοντος, αλλά η συνεργασία στον τομέα ε, των δασών και η εξαγωγή γνώσης και τεχνογνωσία στην δασοκομία είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε τέτοιες σχέσεις και με την Κίνα. Πρέπει να πω ότι μόνο με τον τρόπο αυτό μπορούμε να προωθήσουμε ε, τα πράγματα ε, έτσι ώστε και στην Κίνα να επιτύχουν και εκείνοι τους στόχους τους. Έχουμε ε, καλούς και κοινού στόχους, πάντως είναι γεγονός ότι χρειάζονται και την βοήθεια των άλλων χωρών. Άρα εδώ απαιτείται διεθνής συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Νομίζω ότι καταλάβαμε ποιες είναι οι προτεραιότητές σας και ε, καταλάβατε κι εσείς ποιες είναι οι δικές μας ε, προτεραιότητες. Έχουμε έξι ή μάλλον πέντε μήνες ακόμα στην διάθεσή μας για να έχουμε μια καλή και στενή συνεργασία και σίγουρα θα έχουμε ξανά την ευκαιρία ε, πριν από την, ε, το τέλος της Προεδρίας σας, ε, ελπίζουμε τουλάχιστον να έχουμε την ευκαιρία να σας ξαναδούμε, να μας πείτε τι γίνεται και με τι θα έχει γίνει με τις διαδικασίες που αφορούν το ΠΔΠ και την ΕΚΑΠ που θα έχουν ολοκληρωθεί. Πολύ ωραία, ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα όλη αυτή η συζήτηση. Θα κάνουμε ένα πολύ μικρό διάλειμμα και μετά θα συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα θέματα της ημερησίας διατάξεων.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 Item. Λοιπόν, πρόεδρος, έγκριση ημερησίας διατάξεως, δύσκολα πράγματα αυτά. Αλλά νομίζω ότι τα καταφέραμε, εγκρίναμε τη μέρησια διάταξη. Μπορούμε να περάσουμε στο δεύτερο σημείο λοιπόν. Ε, μερικές ε, ανακοινώσεις έτσι χρηστικές. να υπενθυμίσω κάποιους ε, κανόνες, μια και είναι η πρώτη συνεδρίαση που έχουμε σήμερα. Μήπως θα μπορούσατε λίγο, εάν ε, δεν ε, σας ενδιαφέρει το θέμα, να μην κάνετε πηγαδάκια και να εγκαταλείψετε την αίθουσα, λέει ο Πρόεδρος. Thank you. So the first uh, information to be shared is that the interpretation is available. Uh, λοιπόν, έχουμε διερμηνία σε 20 ε, γλώσσες. Η γραμματεία όμως μας είπε το εξής, εάν ξέρετε ότι έχετε ζητήσει διερμηνία προς τη γλώσσα σας, αλλά γνωρίζετε ότι δεν πρόκειται να παρακολουθήσετε την συνεδρίαση, να το λέτε έτσι ώστε να μειωθούν τα έξοδα της διερμηνίας. Νομίζω ότι αυτό σημαίνει καλύτερη διαχείριση πόρων, πράγμα που συμμεριζόμαστε όλοι. Γιατί όλοι άλλωστε είμαστε φορολογούμενοι πολίτες και πληρώνουμε ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Of good management of... Άρα ε, καλή χρήση των ε, πόρων. Επίσης, όσον αφορά το χαρτί, Ηλεκτρονικά θα είναι τα έγγραφα στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, άρα καλή διαχείριση και των ε, άλλων πόρων πλην των δημοσιονομικών που ανέφερα προηγουμένως. Υπάρχει και η application ή e meeting, ε, δεν ξέρω αν θέλει η γραμματεία να δώσει περισσότερες πληροφορίες, όχι. Εν πάση περιπτώσει, εάν έχετε οποιαδήποτε ανάγκη περαιτέρω πληροφορία όσον αφορά το θέμα αυτό, απευθύνεστε στη γραμματεία. Τρίτο σημείο, χρηστικό πάντα. Θα έχετε λάβει φαντάζομαι ήδη ε, στα έγγραφά σας αυτή την επιστολή Welcome Back. Το Welcome Back, αυτή τη δέσμη των μέτρων, των ε, εγγράφων, συγγνώμη. Εάν έχετε πάντως ερωτήσεις, παρακαλώ. Τέταρτο. Mm έχει αλλάξει και η γραμματεία, τα πρόσωπα της γραμματείας δηλαδή. Είμαστε πολύ τυχεροί γιατί έχουμε την κυρία Σαραμπλό, επικεφαλής της ομάδας, της μονάδας αυτής. Έχουμε δουλέψει μαζί την ε, προηγούμενη εβδομάδα και είναι πραγματικά πολύ αποτελεσματική. Νομίζω ότι έχουμε εμείς την μεγαλύτερη γραμματιακή μονάδα, ομάδα υποστήριξης, ε, 28 άτομα ε, και εν πάση περιπτώσει είτε είστε εισηγητής, είτε σκιώδης, είτε έχετε οποιαδήποτε ε, ερώτηση, μη διστάσετε. Uh, it's very, very helpful uh, to have Sarah and uh, her team. Ωραία λοιπόν, το λύσαμε και αυτό. Τελευταία πληροφορία. Η Τίνα Ζιζαρέβιτς έφυγε μετά από 7 χρόνια πιστής ε, ε, γραμματιακής υποστήριξης ε, στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και της ευχόμαστε καλή τύχη όπου και αν έχει πάει. Αύριο θα έχουμε πολιτικά πιο ευαίσθητα θέματα να συζητήσουμε. Θα συζητήσουμε και για την ΚΑΠ, θα συζητήσουμε για πολλά θέματα. Λοιπόν, τελευταίο σημείο της ημερησίας διατάξεως τώρα Γενικός Προϋπολογισμός Ευρωπαϊκής Ένωση για το οικονομικό έτος 20 και θα σας τα πω στα γαλλικά, αν δεν διαφωνείτε με αυτήν την καινοτομία μου. Εγώ ως πρόεδρος τούτη της Επιτροπής ορίστηκα από τους συντονιστές ως εισηγητής για αυτήν την γνωμοδότηση επί της, ε, του προϋπολογισμού ως ήθιστε κάθε έτος. Θα συμμεριστώ λοιπόν μαζί σας ως ε, εισηγητής και συγγραφέας του κειμένου κάποια στοιχεία ε, τα οποία περιλαμβάνονται στο έγγραφο το οποίο θα μεταβιβάσουμε, θα δώσουμε στην Κομισιόνα. Το πρώτο μήνυμα το οποίο θέλουμε να περάσουμε είναι το εξής το κατόφλι του 20% δαπανών για το κλίμα, που είναι στόχος του παρόντος ΠΙΔΕΛΤΑΠΗ, δεν επετεύχθη. Μια και Μέχρι τώρα οι δαπάνες ε, για το κλίμα είναι της τάξης του 19,7%. Κοντεύουμε στο 20% αλλά ε, εμείς θα θέλαμε να το έχουμε ξεπεράσει λίγο το 20% παρά να βρισκόμαστε ακόμα πιο κάτω. Ζητούμε λοιπόν ε, την τελευταία χρονιά του παρόντος πιδελταπή να έχουμε μια επιτάχυνση των διαδικασιών που αφορούν το κλίμα έτσι ώστε να μπορέσουμε να επιτύχουμε τον αρχικό στόχο στόχο του 20%. Δεύτερο σημαντικό στοιχείο που θα περιλαμβάνεται είναι το εξή. Στη συζήτηση ε, στο Συμβούλιο που έδωσε την θέση του την 11η Ιουλίου, οι δαπάνες που αφορούν το πεδίο ελέγχου ε, της Επιτροπής μας ε, περικόπησαν κατά 1,5 δις ε, ευρώ. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν στις συζητήσεις που θα έχουμε και με την Κομισιόν και με τους Υπουργούς να περάσουμε ξεκάθαρα το μήνυμα ότι εμείς θα επανυποβάλλουμε τροπολογίες έτσι ώστε αυτό το 1,5 δις δαπανών υπέρ του περιβάλλοντος που περικόπησαν να ξαναεισαχθούν στον προϋπολογισμό 2020. Θα υπάρχουν και κάποιοι και άλλα στοιχεία της γνωμοδότησης τα οποία δεν θα αναφέρω τώρα για να φτάσω σε κάτι σημαντικό. Είναι σημαντικό και άλλωστε το υπενθύμησε και ο Υπουργός πριν από λίγο οι υπηρεσίες, ε, οι οργανισμοί ε, που βρίσκονται στο πεδίο επίβλεψης της Επιτροπής μας να έχουν τους πόρους που είναι απαραίτητοι έτσι ώστε με πλήρη ανεξαρτησία ε, να εφαρμόσουν ε, τις, ε, την εργασία τους, να υλοποιήσουν την εργασία τους. Να υπάρξει λοιπόν και οικονομική αλλά και επιστημονική ανεξαρτησία. Αυτό είναι κάτι απαραίτητο και θα πρέπει να υπογραμμιστεί στην παρουσίαση του προϋπολογισμού 2020 που θα πρέπει να είναι στο ύψος των αναγκών και των φιλοδοξιών των υπηρεσιών αυτών. Τελευταίο στοιχείο του οποίου θέλω να επιμείνω. Αυτός ο προπολογισμό είναι ο τελευταίος του ισχύοντος πι Άρα, θα πρέπει ήδη να μεταφέρουμε εμείς ως βουλευτές ε, και να ζητήσουμε από την ε, Κομισιόν ε, να μεταφέρει ο προπολογισμό αυτός κάποιες αρχές οι οποίες αναφέρθηκαν και από τη νέα Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θέλουμε λοιπόν ε, να αναφέρεται, να καταδεικνύεται σαφώς η νέα κατεύθυνση ε, που δίνει η νέα πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έτσι όπως μας την ανέφερε τουλάχιστον στο Στρασβούργο, για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Ε, επίσης, προβληματισμός σε σχέση με την γενική ευθυγράμμιση του προϋπολογισμού πέριξε τη Συμφωνία των Παρισίων και βάση και των συζητήσεων με τον ΟΣΑ. Μέχρι τώρα δεν έχουν ληφθεί ληφθεί σοβαρά και επαρκώς υπόψη τα στοιχεία αυτά. Θα θέλαμε τώρα να ε, είμαστε βέβαιοι ότι θα συμπεριληφθούν. Αυτά είναι εντάχει κάποια από τα στοιχεία τα οποία ήθελα να μοιραστώ μαζί σας, μια και θα είμαι ο εισηγητή ε, ε, της γνωμοδότησης αυτής. Τώρα θα ξαναβάλω το καπέλο του Προέδρου, θα τα πω αγγλικά γιατί ω προέδρο πρέπει να τα λέω αγγλικά. Miss Ευχαριστώ πολύ. Εγώ εκπροσωπώ την κυρία Βαλεάν, την σκιώδη ε, εισηγήτρια εκ μέρους του ΕΛΚ. κυρία Βαλεάν όμω ε, είχε κάποιε συναντήσει τώρα για την αυριανή συνεδρίαση τη Επιτροπής Ήτρε. Θεωρεί λοιπόν, κυρία Βαλεάν, ότι ιδίω στο τελευταίο έτο του ΠΔΕΛΤΑΠΗ θα πρέπει να υπάρξει ένα φιλόδοξο προπολογισμό για την κλιματική δράση και το σχετικό πρόγραμμα για την προστασία της βιοπικιλότητας. Είναι αναγκαίο αυτό ε, ως γέφυρα και προς το επόμενο πι που από ό,τι αναμένεται θα έχει χαμηλούς ρυθμούς εκκίνησης μέχρι ότου καταστεί επιχειρησιακό. Ακούσαμε τις κατηδίες γραμμές από την Ursula von der Leyen. Χρειάζεται επιτάχυνση ε, στο στόχο της μείωσης των εκπομπών. Άρα θα πρέπει να ενισχύσουμε τη μετάβαση ε, από τον άνθρακα στο φυσικό αέριο, μεταξύ άλλων. Θα πρέπει λοιπόν ε, για την κατάρριση του προπολογισμού να εστιάσουμε στις νέες προτεραιότητες. Ευχαριστώ. Σοσιαλιστέ Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ποιος είναι εκπρόσωπός σας? Εσείς. Δεν είναι εδώ ο σκιώδης μας, λέει η κυρία Σαλντεμός. Δεν μπορούμε να πούμε πολλά λοιπόν. Πέραν τούτου θα υποστηρίξουμε την προσπάθεια να αλλάξει μεγαλύτερη χρηματοδότηση για τους εκτελεστικούς οργανισμούς ώστε να είναι εξασφαλισμένη η ανεξαρτησία τους. Ευχαριστώ. Πρόεδρος μέσω των Πρασίνων. Βλέπω τον Πασέικ Χάουτ. Όχι, δεν τον βλέπω. Δεν μιλάει κανείς για να πει τίποτα για τον προπολογισμό της ΕΝΒΙ από τους πράσινους. Να καταγραφεί αυτό. IND. Δεν έχω κάποιο όνομα. Είσαι άρα, κυρία Ζαλίας, για τρίτη φορά παίρνετε το λόγο σήμερα. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Να πω καταρχάς ότι συμφωνώ απόλυτα με τον Πρόεδρο. ότι ναι, αυτό το ποσό που αναφέρατε ίσως να μην είναι υπερβολικό, αλλά αν δει κανεί για πόσα χρήματα μιλάμε στην πράξη, δεν είναι και εύκολα να βρεθούν. Πρέπει λοιπόν να τα διεκδικήσουμε αυτά τα χρήματα και να διαρωτηθούμε γιατί ε, παρέμεινε ανεκμετάλλευτο το κονδύλι αυτό και γιατί αυτό είχε ως αποτέλεσμα τις μελικές περικοπές. Συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπατε. Και μάλιστα εμείς με τροπολογία μας ζητάμε και κάτι ακόμη περισσότερο. Καθότι αυτό θα είναι και αφετηρία της συζήτησης για τις μελλοντικέ δημοσιονομικές προοπτικές. Θέλουμε λοιπόν να επιστήσουμε την προσοχή σας σε ένα διαφορετικό ζήτημα για το 3 συγκεκριμένα, όπου προτείνουμε μια τροπολογία. Θέλουμε ένα ευρωπαϊκό Green Deal μια πράσινη ε, συμφωνία ε, που φαίνεται να είναι στα σχέδια της νέας Προέδρου της Κομισιόν. Δεν υπάρχει όμως κάποιο κάποια νομική βάση, δηλαδή δεν έχουμε στα χέρια μας κάτι απτό μέχρι στιγμής. Οπότε δεν μπορούμε σε τέτοιες ιδέες ε, αόριστες, όσο ωραίες και ανακούγονται, δεν μπορούμε να βάλουμε κάποια συγκεκριμένα κονδύλια να τα συσχετίσουμε αυτά, θα τα πούμε και στις τροπολογίες μας. Οι προκατοχοί μας ανέλαβαν κάποιες δεσμεύσει. σε ό,τι αφορά τον ασμό φαρμάκων, τον οργανισμό πρόληψης ενώσεων κτλ. Περισσότερα μέσα και κονδύλια πρέπει να δοθούν για περισσότερες αρμοδιότητες. Αν λοιπόν ανέλαβαν αυτή την ευθύνη οι προκάτοχοί μας, νομίζω ότι και εμείς πρέπει να πράξουμε αναλόγως, ώστε εκτελεστικοί αυτοί οι οργανισμοί να έχουν στη διάθεσή τους περισσότερα μέσα για να μπορέσουν να φέρουν πέρα στα καθήκοντά τους, που είναι περισσότερο. Ευχαριστώ. Από την Κούε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εμείς είμαστε ικανοποιημένοι με το σχέδιο της Προεδρίας για τα πιο σημαντικά στοιχεία τουλάχιστον που μας απασχολούν αυτά περιλαμβάνονται. Άλλος κανείς θέλει το λόγο, κάποιο ερώτημα, κάποιο σχόλιο, όχι. Μάλιστα. Θα δώσω τώρα το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο Ζήλ Ζοντελέ πρώτα από την DG Move. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και συγχαρητήρια για τα νέα σας καθήκοντα στην Επιτροπή ΕΝΒΗ. Εμείς ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ακούσαμε στην πραγματικότητα ερωτήσεις επί του προπολογισμού, οπότε δεν έχω και να απαντήσω σε κάτι. Ε, βεβαίως ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει γνώση και είναι θετικά διακείμενη στα σχόλια που ακούστηκαν. Όπως ξέρετε είναι το τελευταίο έτος εφαρμογής ε, ε, του δημοσιονομικού πλαισίου. Τα προγράμματα λοιπόν αυτή τη στιγμή είναι στο πιο στο φόρτε τους ας πούμε ε, ιδιαίτερα στο ό,τι της πληρωμές υπάρχουν μια σειρά από δείκτες που δείχνουν ότι τα προγράμματα που είναι εξελίξη όπως το πρόγραμμα LIFE ε, φέρνουν αποτέλεσμα για τη συντήρηση των ειδών ε, ε, για την προστασία των βιοτόπων, στην, τη μείωση των εκπομπών αλλά και τη μείωση των αποβλήτων. Ε, ένα-δύο σχόλια μετά τις παρεμβάσεις των βουλευτών. Θα ήθελα να πω πρώτα απ' όλα ότι βεβαίω είμαστε μόλις το 19,7% ό,τι αφορά τη συμπερίληψη του κλίματος στο σύνολο των δραστηριοτήτων που έχουν να κάνουν με τις δαπάνες και συμφωνούμε ότι δεν αρκεί αυτό το ποσοστό όμως, εάν δούμε την εξέλιξη τα τελευταία έτη, η τάση είναι ενθαρρυντική. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να χαλαρώσουμε. Συμφωνώ απόλυτα με τον Πρόεδρο. Καλύτερα να ανέβουμε κι άλλο παρά να μείνουμε στάσιμοι ή να κατέβουμε. Ε, πάντως πάμε προς την κατεύθυνση. Δεύτερον, είμαστε σε μια κάπως δύσκολη περίοδο όπως γνωρίζετε, διότι από την 1η Νοεμβρίου προβλέπεται ένα κράτος μέλος ε, να αποχωρήσει από την Ένωση και αυτό αντιλαμβάνεστε ότι έχει επιπτώσεις. Ε, για τον προπολογισμό του 2020 δεν θα υπάρξουν κάποια μεγάλα προβλήματα, αλλά στα πλαίσια των συζητήσεων για την ερχόμενη περίοδο θα πρέπει και αυτό να το λάβουμε υπόψη μας. Μεταξύ των θεμάτων που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι επίσης τις συζητήσεις ε, στο Πουδουπού υπάρχει το θέμα των υπηρεσιών, των οργανισμών, το ανέφεραν δύο μέλη εδώ είναι κάτι που δείχνει ότι έχουμε αυτόν τον συνολικό προπολογισμό για αυτού του οργανισμού του αποκεντρωμένου, που υποστηρίζει αυτού του οργανισμού, ε, υποστηρίζει την Κομισιόν ε, και την Ευρωπαϊκή Ένωση για του στόχου που έχουμε θέσει. Υπάρχει ένα ζήτημα ουσία όμω. Ε, όταν προκύπτουν νέα καθήκοντα μετά από συναπόφαση, συχνά ο, δεν προβλέπεται και ο αντίστοιχο προπολογισμό. Είναι σημαντικό λοιπόν στην επόμενη θητεία, πέρα από το συνολικό προπολογισμό που διαπραγματευόμαστε, να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις διάφορες διαπραγματεύσεις που γίνονται ε, γύρω από τα διάφορα νομοθετήματα, όταν προκύπτουν κάποια νέα καθήκοντα για τους οργανισμούς, ο επιπλέον προϋπολογισμός, οι επιπλέον πόροι, ε, οι ανάλογοι, ε, να προβλεφθούν σε αυτή την απόφαση. Μια και είναι η πρώτη συνάντηση πάντως της Επιτροπής αυτής με τη νέα τη σύνθεση. Ήθελα να σας πω ότι η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος, αλλά και η Γενική Διεύθυνση Κλίμα και η Γενική Διεύθυνση Υγείας, ε, προφανώς και είμαστε στην ε, διάθεσή σας να συζητήσουμε με τη γραμματεία της Επιτροπής ΕΝΒΗ, αλλά και για όλες αυτές τις πτυχές να συζητήσουμε, να δώσουμε περισσότερο πληροφορίες που ενδεχομένως να σας λείπουν. Ε, και αν έχετε και άλλες ερωτήσεις, οι συνάδελφοι από τη Διεύθυνση υγείας ή κλίματος είναι στη διάθεσή για να απαντήσουν. Ευχαριστώ πολύ. Να δώσω τώρα το λόγο στον εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης Κλίμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να σας συγχαρώ ε, για τα νέα σας καθήκοντα. Απάντησε ήδη ο συνάδελφος ε, εν μέρη στο θέμα του climate mainstreaming. Υπάρχει μια θετική τάση βεβαίως. Το γεγονός ότι δεν φτάσαμε στο 20% είναι επειδή στην αρχή ουσιαστικά είχαμε πολλά προβλήματα. Το 2014 το 2015 ε, ήμασταν πολύ πιο κάτω. Έξω Έκτοτε όμως έχουμε καλύψει το χαμένο έδαφος, έχουμε φτάσει στο 19,7% μέσο όρο τώρα, δεν είναι τόσο άσχημα τα πράγματα διότι βασιζόμαστε στο σχέδιο προπολογισμού, έτσι. Μπορεί τελικά μάλιστα να είμαστε πάνω από το ποσοστό αυτό. Βεβαίως ε, το σχέδιο γνωμοδότησή σα ε, το βρίσκουμε ποσοστό, ιδιαίτερα το σημείο 1, πρέπει να είμαστε πιο φιλόδοξοι για το μέλλον. Και αυτό ευθυγραμμίζεται με αυτό που ε, είπε ο Γενικός Διευθυντής μας. Στην παρούσα πρόταση για το επόμενο πολιτισμό δημοσιονομικό πλαίσιο, η Κομισιόν ε, είχε ζητήσει 25% climate mainstreaming. Ε, κατά τα λοιπά, εξετάζουμε πώ μπορούμε να κάνουμε περισσότερα. Είναι πολλά τα ζητήματα επιτάπητο. Ε, όλα τα κονδύλια που θα χρειαστούν για το ε, νέο deal για την Ευρώπη η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων που θα μπορούσε να μετατραπεί μέρος σε κλιματική τράπεζα. Ε, μιλάμε για ένα τρισεκατομμύριο, ε, ένα τρισεκατομμύριο επενδύσεις που, που για την επόμενη δεκαετία η νέα πρόεδρο της Επιτροπής. Είναι τεράστια η πρόκληση. Θα πρέπει λοιπόν να ενώσουμε τις δυνάμεις μας στην Κομισιόν, στο Κοινοβούλιο για να τα καταφέρουμε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Θα δώσω τώρα το λόγο στον τελευταίο εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Γενική Διεύθυνση Υγείας, σαν τε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν θα επαναλάβω αυτά που είπαν οι συνάδελφοι για το τελευταίο έτος του πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου. Ένα σημαντικό όμω σημείο στο σχέδιο κειμένου σας για την ΕΦΣΑ. Ε, για την ΕΦΣΑ όντως υπάρχει μια σημαντική αύξηση προσωπικού που ανταποκρίνεται και στην οικονομική δήλωση που συνοδεύει το, την νομοθεσία Food Law. Κατά τα λοιπά, ε, βεβαίως καλωσορίζουμε την πρόθεση της Επιτροπής Ένβη ε, να εγκρίνεται το σχέδιο προβλογισμού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Okay, thank you. Σας ευχαριστώ πολύ. πέραν τώρα του πεδίου αυτή τη νομοδότηση, καλό θα ήταν ίσω σε κάποιο μεταγενέστερο στάδιο να γίνει μια συζήτηση εδώ για το τι σημαίνει ε, η ευθυγράμμιση με τη Συμφωνία των Παρισίων για τον προπολογισμό. Είναι μια διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη με ορισμένα κράτη εκτό και εντό Ένωση. Και καλό θα ήταν να ακούσουμε και τι δικέ σα απόψει για να ξέρουμε τι αυτό συνεπάγεται για το πολιετές. Δεν μιλάμε για ένα νούμερο συγκεκριμένο, θα είναι 20, αν θα είναι 25, πάνω από 25 μέχρι το 2030, γενικώ για τον προπολογισμό και πώς αυτός θα διαμορφωθεί. Θα επανέλθουμε σε αυτό το χρόνο. Λοιπόν, προθεσμία κατάθεση τροπολογιών, εφόσον και έχετε να καταθέσετε τροπολογίες, αύριο, 3 το μεσημέρι, λίγη προθεσμία και θα επανέλθουμε στην Επιτροπή μας 4 Σεπτεμβρίου θα ψηφίσουμε και θα πω και τα υπόλοιπα βήματα μέχρι να φτάσουμε στην ψόφαρη στην Ολομέλεια. Νομίζω ότι εδώ ολοκληρώθηκε η ημερήσια διάταξη για σήμερα. Αύριο συνεδριάζουμε ξανά στις 9 και 30, όχι 9, παρακαλώ σημειώστε το, 9 και μισή το πρωί. Θα τα πούμε αύριο.